Οι πράξει που εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 78. Δημοσιεύονται επίση. Να περάσουμε στο σχέδιο. Στο... Ο κύριο Βέμπερ έχει λόγο για, το... για την ε, μερίσια διαταξή. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να ασχοληθούμε με την κατάσταση στη Ρουμανία τις επόμενες ημέρες. Έγιναν επίσημες έρευνες της εισαγγελία κατά του ε, Πρωθυπουργού Σέφα και ο κύριος Πόντα κατηγορείται για 17 ζητήματα και οι σοσιαλιστές ε, στο Κοινοβούλιο της Ρωμανίας μπλοκάρουν ε, την έρευνα των 17 αυτών ζητημάτων παρά το γεγονό ότι ο Φραντ Τίμερμαν, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για τι αρχέ τη εισαγγελία τη Ρουμανία. Σεβόμαστε τα επικυριαρχικά δικαιώματα του Ρουμανικού Κοινοβουλίου, αλλά πιστεύουμε ότι όλοι οι πολίτε περιμένουν και προσδοκούν διερεύνηση των κατηγοριών αυτών. Και επιπρέστατα, η Υπουργό Δικαιοσύνη ε, τη Ρουμανία είπε ότι όλοι όσοι θέλουν να βγουν να διαδηλώσουν στου δρόμου, ε, θα διωχθούν, θα συλληφθούν ενδεχομένω. Πρόκειται για κάτι απαράδεκτο από πλευρά ε, του κόμματο του ΕΛΚ. Για τέτοιο περιορισμό μιλάμε του δικαιώματο αυτού του σημαντικού της ελευθερίας έκφρασης. Θα πρέπει και της διαδήλωσης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και θα πρέπει να το συζητήσει και ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Εμείς ως ΕΛΚ ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω διαφορετικά νέα από αυτά που μόλις ανέφερε ο συνάδελφος Βέμπερ. Τουλάχιστον το τελευταίο τμήμα της παρέμβασής του. Ωστόσο, εμείς οι σοσιαλιστές συμφωνούμε ότι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών καθώ και στην τακτική διαδικασία του Κοινοβουλίου, όπω έχουμε κάνει και σε άλλε περιπτώσει. Συμμεριζόμαστε το γεγονό ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με την αποκλειστική ε, βάση των ε, πραγματικών γεγονότων. Η αρχή που θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά όλων των δημοκρατικών θεσμών είναι το τεκμήριο αθεότητας και θα πρέπει να βασιστούμε καταρχάς σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, έχω διάφορους συναδέλφους πριν τον το λόγο, αλλά τώρα συζητάμε την ε, ε, ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, όχι της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι μου δίνεται η εντύπωση από τους ομιλητές του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών ότι θα πρέπει να παρακαλώσουμε την Επιτροπή Κοινωνικών Πολιτικών Ελευθεριών να το κοιτάξει το θέμα. Γι' αυτό θα παρακαλέσω τον συνάδελφο Μωράες ε, να το αναλάβει και να το βάλει στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Η κυρία Χάρμς ζήτησε το λόγο. Παρά το γεγονός ότι διακρίνω τη συνένεση των δύο ομάδων, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συνειδητήσουμε στην διάσκεψη των προέδρων. Και τέτοια θέματα σε κανονικέ συνθήκε μπορούμε να τα κοιτάμε στην διάσκεψη των Προέδρων. Σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό επιπρόσθετα, κυρία Αρχάμ, λέει ο Πρόεδρο, αλλά εξ όσων κατάλαβα από του συναδέλφου μου, ζήτησαν να ασχοληθεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών το θέμα αυτό. Μπορούμε παρόλα αυτά να το συζητήσουμε στη διάσκεψη των Προέδρων την Πέμπτη. Κανένα πρόβλημα. Αχα, Μάλιστα, πολύ ωραία. Προτού θεωρήσετε ότι θεωρήσετε ότι είστε ενοχλημένοι, να πω ότι θα κάνουμε και τα δύο. Θα το βάλουμε και στην διασκέψη των Προέδρων και την... θα μπει στην Επιτροπή στην ατζέντα της Επιτροπής. Όχι, δεν μπορώ να δεχτώ τώρα άλλε παρεμβάσει για το θέμα αυτό. Για κάποιο άλλο θέμα θέλετε, κύριε Γιούρεκ, το λόγο, εάν θέλετε το λόγο για κάποιο άλλο θέμα, μάλιστα. Κάτι διαφορετικό αλλά παρόμοιο, πρόεδρε. Πριν από ένα μήνα είχαμε ένα δημοψήφισμα στην Ιρλανδία και ένας νέος ορισμός για το τι είναι η οικογένεια ε, προβλέφθηκε για το σύνταγμά μας. Βέβαια υπήρξαν κάποιες αμφιβολίες και αμφισβητήσεις για το πώς διεξάχθηκε η εκστρατεία, η ενημερωτική εκστρατεία για το δημοσίευμα αυτό και μάθαμε ότι η χρηματοδότηση της εκστρατείας αυτής ξεκίνησε από κρατικούς θεσμούς οι οποίοι απείλησαν πολιτικούς να τους περιθωριοποιήσουν Είμαστε στην Ολομέλεια της, ε, στην, στην ατζέντα της Ολομέλειας, στην μερίσια διάταξη της Ολομέλειας. Αν θέλετε να ζητήσετε το λόγο για κάποιο άλλο θέμα, πρέπει να το ζητήσετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε γενικές δηλώσεις αυτή τη στιγμή και παρεμβάσεις. Naruszone zostały fundamentalne zasady demokratyczne, w tym przede wszystkim zasada tej Πρόκειται για μια πρώτη μειονότητα η οποία πρέπει να έχει στη δημοσιότητα τα ίδια δικαιώματα και γι' αυτό λοιπόν ζητώ να συζητηθεί το δημοψήφισμα λοιπόν. Το θέμα είναι κατά πόσον έχουν και είχαν και οι δύο πλευρές το δικαίωμα και τις ίσες ευκαιρίες να εκπροσωπηθούν. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, για την ημερήσια διάταξη δεν βλέπω να υπάρχουν σήμερα ε, αιτήματα. Για την Τρίτη, η έκθεση Κονφεράτη ζητήθηκε να αναβληθεί για τον Ιούλιο και να συζητήσουμε την έκθεση Λαντσπέρκης για τις ε, σχέσεις ε, με τη Ρωσία που είχε προβλεφθεί για την Τετάρτη. Κύριε κύριο Σαλόμ ζήτησε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την έκθεση που φέρει το όνομα του κύριου Κοφεράτη. Είναι μια σημαντική έκθεση Υπάρχουν κάποια ζητήματα σοβαρά, από των οποίων όμως δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Υπάρχει δυνατότητα επίτευξης βέβαια της συμφωνίας αυτής, αν υπάρξει λίγο περισσότερος χρόνος και αν ξεκινήσει διαβουλεύσει ο κύριο Κοφεράτη με τι διάφορε πολιτικέ ομάδε. Θα ζητούσα λοιπόν εξ ονόματο τη δική μου πολιτική ομάδα ε, να αναβληθεί, να καθυστερήσει και να πάει τον Ιούλιο η συζήτηση και η ψήφιση τη εκθέσεω για να έχει το χρόνο αυτό ο κύριο Κοφεράτη. Ποιο είναι υπέρ του αιτήματο αυτού και θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε και η ομάδα της GUE NGL θεωρεί ότι είναι καλύτερα να υπάρξει μια μικρή αναβολή για την συνεδρίαση του Ιουλίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με περισσότερη οριμότητα και ετοιμότητα το θέμα αυτό, το οποίο πραγματικά έχει μεγάλη σημασία. Δεν πρέπει να βιαστούμε. Ποιο θα ήθελα να μιλήσει κατά του αιτήματο αυτού. Κανείς. Ας ψηφίσουμε λοιπόν το αίτημα αναβολής του κυρίου Γκερέρο. Ποιο είναι υπέρ της αναβολής. Ποιο είναι κατά. Άποχες. Εγκρίνεται λοιπόν. Η έκθεση Κομφεράτη θα αναβληθεί για μετέπειτα, σε μετέπειτα σύνοδο. Την ε, Τρίτη το πρωί θα συζητηθεί η έκθεση Λανσμπεργκής. Για την Τετάρτη τώρα. Το EFTD, η ομάδα του EFTD να συζητηθεί και να συνεχιστεί η, έκθεση, η συζήτηση για την έκθεση Λάνια για το TTIP. Ο συνάδελφος Άρνοτ παίρνει το λόγο για να δικαιολογήσει το αίτημα αυτό. Uh, yes, Mr. President, uh, the reason for this is... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο λόγος είναι πολύ απλό. Σε 24 ώρε, σε μια από τις ε, μικρότερε περιοχέ των εκλογικών μας περιφερειών, χίλια άτομα ήρθαν σε επαφή μαζί μου για να ενημερώσουν, ε, για να μου ζητήσουν να παρέμβω. Ε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ και πρέπει τα θέματα αυτά να μας αποσχολήσουν και να συζητηθούν. Δεν νομίζω ότι θα είναι δίκαιο στην, για την εταιρική σχέση, τη διατλαντική εταιρική σχέση, να μην το προβλέψουμε. Έχουμε πολλές, πολλά αιτήματα χρονογόρευσης από πολλά μέλη αυτής της ομάδας. Ε, οπότε καλό είναι να δείξουμε και στο κοινό μας την, την γνώμη ότι μας ενδιαφέρει αυτό. Θα πρέπει δηλαδή η έκθεση αυτή να δείξουμε ότι μας απασχολεί και την εξετάζουμε σοβαρά. Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο αυτού. Υπέρ του αιτήματο Άρνοτ. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο κατά του αιτήματο. Κατά, κύριε Γερέρο. Ακούστε. Δεν είμαι ακριβώς κατά. Απλά αυτό αυτό Γελάστε, γελάστε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να αποφύγουμε είναι να μην γίνει η ψηφοφορία την Τετάρτη. Τι θέλω να πω. Εάν παραταθεί ε, για το απόγευμα η συζήτηση, θα πρέπει να ψηφιστεί την πέμπτη έκθεση. Είμαι υπέρ, η ομάδα μου τουλάχιστον είναι υπέρ του να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αλλά εγώ έλεγα ότι αυτό μπορεί να γίνει εάν δώσουμε περισσότερο χρόνο το πρωί. Αντί να ξεκινήσουμε στις 9, να ξεκινήσουμε στις 8 το πρωί. Δηλαδή να δώσουμε το χρόνο με τον περισσότερο, αλλά το πρωί. Hatte, habe ich gegeben? Kann ja, Herr Kollege, finde. Συνάδελφε, είναι πάρα πολύ ευγενικό που αντιφάστε τόσο άμεσα, κυρία Θα Πάρτε το λόγο, λοιπόν. Is this microphone working now? Yes. We, would be... Δουλεύει το μικρόφωνο. Με τα χαρά να, ξε... να, ζητήσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση νωρίτερα στις 8. Okay. So, da haben wir jetzt Gemeinsamkeit. Μάλιστα, καταλήξαμε λοιπόν σε ένα κοινό το θέλετε να ξεκινήσετε στις 8 και όχι στις 9. Είναι κανείς κατά? Ήθελε να πάρει κανείς το λόγο κατά? της κίνησης των εργασιών στις 8 το πρωί. Μάλιστα. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματο Γκερέρο, να ξεκινήσουμε στις 8, ποιος είναι υπέρ της πρότασης Γκερέρο. Ποιος είναι κατά. Ναι, νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν στις 8 το πρωί την Τετάρτη. Στη συνέχεια, κυρίε και κύριοι, ένα αίτημα των πρασίνων σε ό,τι αφορά το προφορικό ερώτημα για τον αθλητισμό στο Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά και τους αγώνες των Πακού. Οι πράσινοι προτείνουν να υπάρξει ψήφισμα. Η κυρία Λούνατσακ θα πάρει το λόγο για να αιτιολογήσει το αίτημα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, σε οκτώ μέρες οι ευρωπαϊκοί αγώνες θα ξεκινήσουν στον Πακού. Από το περασμένο καλοκαίρι στο Αζερμπαϊτζάν όλοι οι ακτιβιστές ουσιαστικά ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν φυλακιστεί. Και έχουμε ένα προφορικό ερώτημα στην ατζέντα την Τετάρτη το απόγευμα να συζητηθεί. Αλλά δεν ε, συμφωνήσαμε να υπάρξει ψήφισμα. Όλα τα άλλα μεγάλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Μισελ Φόρστ, ε, η δυναμιά το η πρόσωπος του ΑΣΕ για την ελευθερία του τύπου, όλοι έχουν εκφέρει άποψη και έχουν δηλώσει ότι δεν μπορεί στον αθλητισμό να αγνοούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω λοιπόν ότι όλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα έπρεπε και δεν πρέπει να διστάσει, να κάνει πίσω, θα πρέπει να αρθούμε στο ύψο των περιστάσεων, να αναλάβουμε τι ευθύνε μα και να εκφραστούμε μέσω ενό ψηφίσματο. Θέλουμε ένα σαφέ μήνυμα για να εξασφαλίσουμε ότι άτομα όπω η Λέλα Γιούνο, που ήταν υποψήφια για το βραβείο Ζαχάροφ και πολλοί άλλοι, θα απελευθερωθούν και ότι αυτοί οι αγώνε δεν θα ε, γίνουν υποσκιά τη δύσκολη κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζητώ να υποστηρίξετε το ψήφισμα. Ποιος θέλει να υποστηρίξει την ε, κυρία Λούνατζε και το αίτημά της. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όντω, σε μερικέ μέρε αρχίζουν οι αγώνε στον Πακού. Ο πρόεδρο έχει χρησιμοποιήσει αυτή την εκδήλωση για να προβάλλει αυτά που θέλει σαν βιτρίνα για το καθεστώ του. Όμω είναι ένα καθεστώ απολυταρχικό. Και οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το σύνολο των, ανθρωπίνων, ε, των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα μα το επισημαίνουν αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να μα απασχολήσει τι γίνεται εκεί με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων από τέτοια καθεστώτα. Πρέπει να καταδικάσουμε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Αζερβαϊτζάν. Και όπω το είπε και η κυρία Λούνατσεκ, πρέπει να εκφραστούμε γραπτός. Ιδάλλως δεν έχει την ίδια βαρύτητα η έκφρασή μας. Και γι' αυτό ε, με την ομάδα μας και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ομοφόνος υποστηρίξαμε, ε, όπως και η πράσινη, ότι πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο ψήφισμα. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο για... κατά. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να επισημάνω ότι το θέμα αυτό τέθηκε στην αρμόδια επιτροπή η οποία το απέρριψε και μάλιστα δέχτηκε να γίνει αυτή η συζήτηση διότι η πλειοψηφία της αρμόδιας επιτροπής είπε ότι δεν πρέπει να υπάρξει ψήφισμα. δεύτερον και πιο σημαντικό είχαμε την ευκαιρία και οι συνάδελφοι πριν δεκαπέντε μέρες όταν συζητούσαμε την εταιρική σχέση που είναι πάρα πολύ σημαντική να τεθούν αυτά τα θέματα για το αζερμπαϊτζάν τότε για να έχει τη δυνατότητα και η ηγεσία της ευρωπαϊκής ένωσης και το κοινοβούλιο να θέσει τα ζητήματα αυτά εγκαίρως. δεν τέθηκαν όμως αυτά. τρίτο και επίσης σημαντικό σε είκοσι μέρες γίνεται συζήτηση στο συμβούλιο της ευρώπης για το ζήτημα αυτό όπου εκεί υπάρχει αρμόδια επιτροπή που το έχει εξετάσει. θεωρώ ότι όποιο ψήφισμα σήμερα αποφασίσουμε να υπάρξει δημιουργεί ένα δεδικασμένο και προδιαγράφει τις αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου που είναι το συμβούλιο της ευρώπης. Ε, αυτά τα θέματα πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη όπως επίσης και για την πορεία της εταιρικής σχέσης. άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να εκφραστεί εδώ κατά τη συζήτηση αλλά το να υπάρξει ψήφισμα δεν δίνει το χρόνο σε όλους εμάς να προετοιμαστούμε και να συζητήσουμε και οι πολιτικές ομάδες επίσης να έχουν τις θέσεις τους για να έρθουν οργανωμένα στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ψηφίσουμε την πρόταση της κυρίας Λούνατσεκ. Ποιος είναι υπέρ του ψηφίσματος παρακαλώ. Ποιος είναι κατά. Ποιος απέχει. Απορρίπτεται. Έλεγχος ζητείτε. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εάν ψήφισατε όλοι. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι, λέει ο Πρόεδρος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το έτοιμα. 136 ψήφοι υπέρ, 136 κατά. Τια. Κάτι. Τια. Vielen Dank. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν ε, ο... οριστικοποιείται η ημερήσια διάταξη, το πρόγραμμα εργασιών. Das Αυτό το πρόβλημα το έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Και δυστυχώ δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα εκ των υστέρων. Πολύ ωραία. Κυρία και διαδικαστικό θέλετε να θέσετε. Έχετε το λόγο. Ήθελα μόνο να ρωτήσω, ε, άκουσα ότι κάποιος από τους φιλελεύθερους ε, δεν λειτουργήσε το μηχανάκι του. Η συσκευή ψηφοφορίας. Δεν ξέρω πώς θα ψήφιζε, αλλά αυτό να ληφθεί υπόψη. Είτε ήταν υπέρ, είτε ήταν κατά. Να ληφθεί υπόψη αυτή η ψήφος και ελπίζω να ήταν υπέρ. Θα το λάβουμε υπόψη, λέει ο Πρόεδρο, αλλά γνωρίζετε το πρόβλημα σε ονομαστικέ ψηφοφορίε, σε ηλεκτρονικό έλεγχο ψηφοφορία Κάθε φορά έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Κάποιοι συνάδελφοι βάζουν λάθος τις κάρτες τους, κάποιοι δεν συλλειτουργούν τις συσκευές τους, το γνωρίζω. Πολύ λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω το αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Γι' αυτό λοιπόν ρωτάω διάφορες βορές ψηφίσαν όλοι, όλοι με επικρίνουν κάποιοι μου λένε ότι περιμένω πολύ γιατί θέλω μια συγκεκριμένη ψηφοφορία. Τα ξέρω όλα αυτά, αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να αλλάξει εκ των υστέρων το αποτέλεσμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι οριστικοποιείται το πρόγραμμα εργασιών. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στην έκθεση του κυρίου Ζικέρσκι, ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά το 2015. Το λόγο έχει ο κύριος Ζικέρσκη. ο κύριος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι.